είναι ο καλύτερος τρόπος να ενεργήσουμε. Και θα επιληθούν έτσι όλα τα προβλήματα. Ρίξε το στο γυαλό λοιπόν. Όλα τα προβλήματα, <laughs> εκτός από αυτά τα οποία στοχεύει το θέμα αυτό να λύσει. κυρία Μουσκαρντίνο την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. την ευαισθησία του προβλήματος, την καταδεικνύει η παρουσία του κύριου Επιτρόπου εδώ. Αυτό που μου είναι πιο δύσκολο να καταλάβω σήμερα είναι γιατί δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση του κυρίου Κασπαρή που μου φαίνεται απολύτως νόμιμη και δικαιολογημένη και που εξάλλου επαναλήθηκε και στις επόμενες ε, ομιλίες που ακούσαμε και ερωτήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά κύριε Πίτροπε που το Κοινοβούλιο συνεργάζεται αλληλέγγυα με την Κομισιόν που διάγει μαζί της ε, ένα μεγάλο δρόμο και το Συμβουλίο μας αφήνει ξεκρέμαστους. Τώρα το ερώτημα του μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατή μια δημοσιολάβηση και συγκεκριμένη εργασία είναι απαραίτητη, αναγκαία διότι εάν χρησιμοποιήσουμε λάθος το χρόνο που μας έχουν εκχωρήσει οι πολίτες μας δεν θα δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στις χώρες μας θα χάνουμε το χρόνο μας. Μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Εσείς είπατε κάτι που εγώ υποστηρίζω απόλυτα. Η αμοιβαία ότι ο Πόη δεν ε, πιστεύει στην αμοιβαιότητα κάθε φορά μας κάνει υποσχέσεις και τίποτα δεν τηρείται. Εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Συμφωνούν συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές οικογένειες και σε εποχές κρίσης πρέπει να επιτύχουμε ό,τι είναι δυνατόν για το κοινό καλό της Ευρώπης και των χωρών μας. Ποια είναι λοιπόν η δράση που έχει αναλάβει ο ΠΟΕ, η τα θεσμικά όργανα ενώπιον του ΠΟΕ του ΠΟΕ ώστε η Κίνα μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια να κινηθεί διαφορετικά από ό,τι κινήθηκε σε σχέση με το έστω και ελάχιστο άνοιγμα κάποιας δημόσια σύμβασης. Έγινε κάποια τέτοια κίνηση. Μήπως δεν αληθεύει ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε τις σωστές έκανε μεν σωστέ κινήσει, αλλά με λάθο αποτελέσματα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Δυστυχώ ε, δραματικό, τραγικό. Εμεί ε, δημιουργήσαμε μια διάταξη πληρωμών 30 ημερών. Γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι όσοι έχουν τα μονοπόλια μεγάλης διανομής στην Ευρώπη με αυτή την αιτιολογία της υποχρέωσης των 30 ημερών χαμήλωσαν όλες τις τιμές και απειλούν μάλιστα ότι αν δεν δώσουν με τα χρονολογημένα τιμολόγια θα χάσουν την πώληση εμείς είμαστε κατά του μονοπωλίου, αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν μονοπόλια. Υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι σε κάθε χώρα για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι ένα σπίτι πρέπει να χτίζεται από τα θεμέλια και όχι και από τη σκεπή. Και πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να χτίσουμε αυτά τα θεμέλια και τα τρία θεσμικά όργανα μαζί με, τις, με τους ίδιους λήθους, με τις ίδιες ιδέες ή όχι. Τελευταία ερώτηση. ο κύριος Φρανκ Προύστ. Ναι, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μία σύντομη παρέμβαση. Διότι μπορούμε να διαρωτηθούμε έχουμε την υποχρέωση να καταλήξουμε σε αποτελέσματα διότι το πρόβλημα τέθηκε δεδομένου ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όταν κάναμε ακρόαση σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες κινούνται στην ε, παγκόσμια αγορά, είδαμε ότι υπάρχουν διάφορες ε, δυσλειτουργίες και αν δεν κάνουμε κάτι, όλο και περισσότερο ευρωσκεπτικιστές θα πιστεύουν ότι τα πράγματα λειτουργούν λάθος σε αυτή την Ευρώπη. Όπως έλεγε και ο συνάδελφος ε, δίπλα μου, αυτό το οποίο είναι σημαντικό δεν υπάρχει 6-8, ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, ώστε να δώσουμε προς τα έξω, να στείλει προς τα έξω ένα μήνυμα, λέγοντας ότι η εποχή κατά την οποία η Ευρώπη είχε ανοίξει τις αγορές της χωρίς να υπάρχει καμία αρχή αμοιβαιότητες, παρήλθε. Δεν είμαστε πλέον αφελείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα προς τα έξω. Έχουμε τις ασιατικές χώρες, τις αναδιόμενες, ακόμη και τις είπα, δούμε πώς συμπεριφέρονται, θα πρέπει να ενεργήσουμε, να αντιδράσουμε και να βρούμε τα μέσα που θα μας επιτρέπουν να προστατέψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις θέσεις και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δυσκολίες διείσδυσης σε άλλες αγορές. Ακόμη μία φορά λοιπόν σήμερα Εάν μου επιτρέπετε, θα πω το εξή. Η υποχρέωση που έχουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να προσπαθήσουμε να δούμε την πιο κατάλληλη λύση για να προασπίσουμε τι ε, θέσει εργασίε και τι οικονομία μα γενικότερα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήσει που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ ανοιχτό μαζί σας. Στην αρχή, τέτοιου είδους ασκήσεις δεν μου προκαλούσαν και μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν κινούμε συνήθως σε τέτοιου είδους πλαίσια. Ο Μισελ Μπαρνιέ ήταν μάλλον υπέρ όλης αυτής της ε, διαδικασίε και χρειάστηκε να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση, διότι για πολύ παράξενους λόγους είναι υπεύθυνο για το GPA και εγώ για τις κρατικές προμήθειε τη μερή σχέση. Και λόγω που δεν έχω ακόμη διερευνήσει. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να πω ότι όταν συζητούμε αυτά τα θέματα και όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο έξω, είμαι όλο και περισσότερο πεπισμένος ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους μέσα στη διαθεσή μας. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε συμφωνία με τον Καναδά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν λοιπόν συμφέροντα για τη δική τους αγορά κρατικών προμηθειών η οποία ήταν κλειστή και σε επίπεδο ομοσπονδιακό και σε επίπεδο κάθε ε, περιοχής. Είναι δύσκολα τα πράγματα ότι πρέπει με ένα ομόσπονδο κράτο να συζητήσει τέτοιου είδου θέματα, διότι γίνονται όλα σε δύο επίπεδα και οι συζητήσει πρέπει να γίνουν σε δύο επίπεδα. Και επίσης με την ε, ΣΥΠΑ είναι παραφέρει τα πράγματα σε επίπεδο ΙΠΑ και σε επίπεδο κάθε ποιος χωριστά. Με τον Κανιδά μπορώ να πω ότι είναι καλή συμφωνία και θα είναι πραγματικά μια μεγάλη δυνατότητα ανοίγματος σε αυτές τις χώρες. Αλλά χρειάστηκε να, καταλάβουμε, να καταβάλουμε ένα τίμημα. Δεν μπορούμε να πούμε δεν σας ζητάμε τίποτα γιατί είναι ανοιχτέ οι αγορές. Αυτό που σημαίνει στι διαπραγματεύσει είναι ότι το έχουμε αυτό στη διάθεσή μα και αν το θέλετε θα πρέπει να πληρώσετε. Πρέπει λοιπόν να πω ότι κύριε Φέλνερ, εγώ είμαι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών, είμαι πεπισμένος και είναι λογικό να υπάρχει μια κάποια αμοιβαιότητα. Διαφορετικά πρέπει να, καταλάβ... να καταβάλλετε ένα τίμημα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό κατά την άποψή μου ούτως ή είναι δίκαιο. Απόλυτα. Ένα άλλο ερώτημα που έθεσε. Δεν βλέπω το όνομά σας. Η κυρία Κλάρκιν. τι γίνεται με όλες αυτές τις ε, παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειών αγαθών. Προμήθειας αγαθών. Η πρότασή μας βασίζεται σε ποσοστό ε, ε τοπικού περιεχομένου 50%. Δηλαδή, οποιαδήποτε εταιρεία τρίτης χώρας παραδίδει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αυτό το local content σε ποσοστό 50%. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό σε άλλες περιπτώσεις. Εμείς το έχουμε ορίσει αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, δίδουμε την δυνατότητα να προμηθευόμαστε στα πιο, στις πιο φθηνές αγορές αν θέλετε, υπό τον όρο ότι το ποσοστό δεν θα ε, ξεπερνά το 50%. Γιατί κάπου πρέπει να βάλετε το ορόσημο, το όριο. Τώρα, οι συζητήσεις 47-52% είναι κάτι το γελίο, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ λογικό το 50% το οποίο θεσπίστηκε. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την πρόταση. Βρίσκω ότι είναι πολύ λογική. Ίσως γιατί εγώ την έφτιαξα. Γιατί πιστεύω ότι είναι λογική. Διότι είναι συνδυασμός μιας συνολικής σφαιρικής άποψης και προσέγγισης και προσέγγιση σε ένα ειδικό φάκελο βασίζουμε για το που λέω στο άρθρο 6 κυρίως. Τι λέει το άρθρο 6, διότι πολλοί λένε αφήνεται τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν ή όχι έναν ε, μειοδοτικό διαγωνισμό. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τις αρμόδιες αρχές. Αυτό όμως δεν είναι αληθές. Πρέπει να γίνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να γίνει αυτός ο μυρωτικός διαγωνισμός. Και αυτό το ζήτησαν κάποιοι. Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να δουλεύει, γιατί υπήρχαν τέτοιου αιτήματα. δεν λαμβάνονται μόνοι νομερός κάποιες ε, αποφάσεις. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάποια πράγματα που έχουν αποφασιστεί κοινοτικά ε, εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τους μέσους είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί ερωτηματικά. Λοιπόν, έχουμε αυτή την global approach, αυτή την ειδική προσέγγιση, κάναμε την έρευνα στον σχετικό τομέα και νομίζω ότι το λέει αυτό με σαφήνεια το άρθρο 8 ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να δούμε πώς αντιδρά όλος ο τομέας και να κάνουμε τη σχετική έρευνα να δούμε τι θα ακολουθήσει το δασκαλί και ισορροπημένη λοιπόν είναι η πρόταση πιστεύω διότι από τη μια έχουμε μία προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, με όρια όμως, έτσι. Εάν ε, μία περίπτωση γίνει η γενική τάση, θα πρέπει να την εξετάσει η Επιτροπή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εάν υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα, Φερρυπίν, στην Σλοβακία ή στη Γαλλία, ξαφνικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το απλοστάσιό μας και να απαγορέψουμε τα πάντα. Εμείς ενεργώντας έτσι έχουμε επιτύχει μία ισορροπία. Εάν θέλετε να τα αλλάξουμε και να συζητήσουμε, μπορούμε. Υπάρχει η κατά περίπτωση προσέγγιση και η γενική προσέγγιση. Και εγώ είμαι έτοιμος να εξετάσω ενδεχόμενες τροπολογίες, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι στην έκθεσή σας αν πείτε ότι ε, έτσι έχει η πρότασή σας, αυτές τις τροπολογίες καταθέτουμε και θέλουν να γίνουν οι ΑΒ αλλαγές, έχει καλός. Έχουμε, μέχρι τώρα μας δεν έχουμε πάρει τίποτε από εσάς. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι καινούρια, έχει χρησιμοποιηθεί και στην οδηγία η οποία αφορά τα utilities. To change things. Τις ε, επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Εν πάση περιπτώσει, συζητώντας με τον Μισελ Μπαρνιέ, φτιάχνουμε την πρότασή μα, αλλά κάντε και εσείς που βάλετε τροπολογίες, περιμένουμε την εκθεσή σα. Και κανενό το επιχείρημα δεν υπηρεσχεί σε σχέση με αλλού. Βεβαίω. υπάρχουν κάποιε αρχέ τι οποίε πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τι αρχέ. όχι πάρα πολλέ, βέβαια, διότι αν έχουμε ε, πάρα πολλέ, δυσκολεύεται την κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω ακούσει έως τώρα ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους να μας λέτε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση. Ίσως υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει είμαι διατεθειμένος να ε, συζητήσω αλλαγές και διαφοροποιήσεις μεταξύ του 6 του 8. Ας δούμε πώς διαγράφεται η πλειοψηφία. Αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους μέσα τα χρειαζόμαστε. Και δεν είμαι προστατευτιστής. Μπορείτε να πείτε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί κανεί να πει κανένα ότι εγώ είμαι υπέρ τη προστατευτική προσθήκη. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν έχουμε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αποκλείσουμε κάτι από τι αγορέ μα για θέματα ασφαλεία. Δεν έχουμε καμία τέτοια δυνατότητα, το ξέρετε. Κάποια κράτη-μέλη, ναι. Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε περιπτώσει κρίσιμων βιομηχανιών για εμά θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε κάποια πράγματα. Θα μπορούσα να σα δώσω κάποιο παράδειγμα, αλλά θα το γνωρίζετε ήδη. Δεν μπορούμε να δράσουμε αυτή τη στιγμή. Και ενώ πρέπει να δράσουμε, επειδή πιστεύουμε στι ελεύθερε αγορέ. Δεν πρέπει να είμαστε όμω αφελεί. Έχουμε δικαιώματα και μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα και άλλα πράγματα δεν μπορούμε να τα δεχθούμε. Πρέπει να σας πω ότι το παράδειγμα που θα σας έδινα θα ήταν ιδιαίτερα πιστικό. Αν ήσασταν παρόντες εκεί που το είδα, θα συμφωνούσατε μαζί μου. Πρέπει να πληρώσουμε γιατί είμαστε ανοιχτοί. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Εξαιρετική ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα σας δούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Cristiano, thank you for coming. Αγαπητοί συναδελφοί, έχουμε ακόμη δουλειά πριν τελειώσει αυτή η συνεδρίαση. Είμαστε μια επιτροπή με πολλή δουλειά και πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα, να δώσουμε αποτελέσματα. Ακολουθεί το σημείο 16 τροποποίηση τις οδηγίες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και τις οδηγίες σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή ΕΜΒΗ είναι υπεύθυνη για αυτό το νομοθετικό φάκελο και εμείς είμαστε γνωμοδότες προς την ΕΜΒΗ. Η συγκητής μας είναι ο Ζωζεφ Αντρέας, δεν βρίσκεται εδώ, θα αντικαταστήσει από τον Μπέρντ Λάγκεν. και θα ακολουθήσει τώρα μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Δίνω το λόγο στον Μπέρντ Λάγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη για την Ιωζέφα, δεν μπόρεσε να πάρει το αεροπλάνο και άρα δεν είναι εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο είναι το θέμα μας εδώ. Έχουμε αφενός το ζήτημα της ποσόστοσης βιοκαυσίμων 10% αν θα παραμείνει το ίδιο ή αν θα μειωθεί η Κομισιόν. Προτείνει να το μειώσουμε στο 5% γιατί ε, με λέει πως με την αυξημένη παραγωγή βιοκαυσίμων έχουμε αλλαγή χρήσης γης που αλλιώς θα χρησιμοποιείται για παραγωγή τροφίμων και επίσης έχουμε και τον φόβο πως τα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς δεν έχουν πλέον εκτίματα σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα, αντιθέτως ενισχύονται υπερβολικά. Εγώ θα συμφωνήσω με την Κομισιόν, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πως με τον περιορισμό στο 5% ακυρώνονται πολλές επενδύσεις που έγιναν στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Εάν δεν ακυρώνονται δεν είναι πλέον τόσο συμφέρουσες. Οπότε θα μπορούσε ίσως να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Αλλά γενικά είναι σωστή η προσέγγιση. Μετά υπάρχει μια δεύτερη προσέγγιση ε, να πούμε πως θέλουμε να προωθήσουμε ειδικά τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Δηλαδή, να μην καλλιεργούμε φυτά ειδικά για να γίνουν βιοκαύσιμα, αλλά να έχουμε κάποια υπολείμματα κάποιας άλλης διαδικασίας που θα γίνονται βιοκαύσιμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρξει μια ειδική πιστοποίηση ανάλογα με τη δυναμικότητα που έχουν για τα αερίδια διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά τώρα την πτυχή του εμπορίου, εκεί πέρα έχω σοβαρά προβλήματα. Γιατί βεβαίως εδώ πέρα ενισχύουμε τις εισαγωγές ειδικά όσον αφορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Γιατί αν δούμε πως ήδη και σήμερα έχουμε επιδότηση πάρα πολύ μεγάλη των βιοκαυσίμων. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορούμε να περάσουμε σε αυτή την επιδότηση των εισαγωμένων βιοκαυσίμων χωρίς να υπάρξει κάποια προδιαγραφή όσον αφορά την αηφορία τους. Και κάτι άλλο στην πρόταση της Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε, έχουμε την διπλή ε, αξιολόγηση για τα ε, τα φυτικά, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση μετράνε δύο φορές. Υπάρχει μια διπλή στάθμιση. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης των τιμών είναι απολύτως πιθανόν εισαγόμενα έλεα τηγανίσματος να είναι φτηνότερα από το τοπικό. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή μια τέτοια αγορά Ενό λαδιού τηγανίσματο το οποίο θα έχει χαρακτηριστεί τεχνητά έτσι κιόλας. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε το στόχο μας χωρίς ταυτόχρονα να μειωθεί η παραγωγή τροφίμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, thank you. Next, uh... Η Elizabeth Κόστιγκερ, του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Μπέρντ Λάγκε και την εισηγήτρια. Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε πως ε, τα βιοκαύσιμα πρέπει να παίξουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ειδικά δεδομένης της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Ο Μπερνάγκη ανέφερθηκε στο κριτήριο της αηφορίας, το οποίο λείπει εντελώς. Δηλαδή όταν μιλάμε για βιοκάψιμα, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για τις υπόλοιπες εναλλακτικές. Αυτό το οποίο τίθε λοιπόν με βάση την προσέγγιση της Κομισιόν είναι πού θέλουμε, πως τα πού θέλουμε να κινηθούμε και προς τα δύο καύσιμα βεβαίως και προς τα ανανεώσιμες φύγες ενέργειας. Ή θα επιβαρύνουμε έναν νέο και αναπτυσσόμενο κλάδο στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον Ευρωπαίο παραγωγό, για την ευρωπαϊκή θέση εργασίας. Ο κλάδος αυτός ξεκίνησε από μια α, ρυθμιζόμενη αγορά και έχει νομίζω αντιδράσει σχετικά. Και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική πτυχή στην όλη αυτή συζήτηση είναι όσον αφορά την πρώτη γενιά το τι γίνεται με τις ε, πρωτεΐνες που είναι υψηλής ε, ποιότητας ε, προϊόντα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, ζωοτροφή. Γνωρίζουμε πως στην Ευρώπη εξαρτώμαστε πάρα πολύ από εισαγωγές ζωοτροφών και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό στη συζήτησή μας. Έχουμε και, όπως είπα, την ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή που θα έχουν αυτές οι αποφάσεις ε, στη, στα πρωτεϊνούχα φυτά και τις εισαγωγέ που έρχονται από την Νότια Αμερική εδώ πέρα και τίθεται και το ζήτημα της αηφορίας. Δηλαδή αφενός μιλάμε για την ευρωπαϊκή μας αγορά και από την άλλη λέμε πως ε, εντάξει αν είναι να περάσει τους ωκεανούς για να έρθει στην Ευρώπη, προφανώς δεν είναι και πολύ αηφόρο. Κάτι άλλο σε σχέση με τους παράγοντες ε, αξιολόγησης ε, και οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται εδώ πέρα δεν είναι τόσο απλοί. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που ορίζουν κάποια παραδείγματα, όπου υπάρχουν κάποιες υποθέσεις για το πώς ε, υπολογίζονται αυτοί οι συντελεστές για τις νέες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Αν δείτε, παραδείγματο χάρη, τι γίνεται, σε γενικές γραμμές ε, με την ίδια έκταση είχαμε την διπλάσια ε, παραγωγή. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κάνουμε λανθασμένες υποθέσεις όσον αφορά την ε, πιθανή ε, παραγωγικότητα του ε, εδάφους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αντικειμενικοί και να φροντίσουμε η αλλαγή αυτή τελικά να μην οδηγήσει σε περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να λάβουμε υπόψη και την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών. Έχουμε βέβαια και τις επενδύσεις που ανέφερα ήδη και πρέπει να σκεφτούμε επίσης πως το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η Κομισιόν είναι κάπως περιορισμένο. Οι επιχειρήσει οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με μια έτσι πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση. Όσον αφορά δε, τα βιοκαύσιμα τρίτη γενιά, εδώ πέρα συμφωνούμε, όπω και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Πρέπει να είναι αυτά τα βασικά σημεία που θα μα απασχολήσουν. Νομίζω πως μπορούμε άρα να συμφωνήσουμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Next. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη σκιώδης, Κατερίνη Γέλντερ από το Άλντε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν έχω να πω ιδιαίτερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γκουε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ζήτημα και η δυστυχή πραγματικότητα είναι ότι οι στόχοι πρασινών μεταφορών για το 2020 έδωσαν κίνητρα για επιζήμια τεχνολογία, ειδικότερα σε βιοκαύσιμα που βασίζονται σε φυτά. Και αν διαβάσετε τα σχέδια δράσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των κρατών, δεν πρόκειται να πλήρουν το στόχο του 10% για τις μεταφορές. Νομίζω ότι είναι σαφές για τα περισσότερα κράτη-μέλη ότι θα το επιτύχουν αυτό μέσω βιοκαυσίμων. Πολλά τα οποία βασίζονται σε φυτά και αυτό θα σημαίνει γενικά μεγάλη αύξηση των βιοκαυσίμων αυτών. Είχε γίνει μια μελέτη νομίζω για την Κομισιόν το 2011 η οποία συμπέρανε ότι τα δύο τρίτα ή περισσότερο κατά τη μετάβαση των, σε βιοκαύσιμα θα έχουν επιρροές ε, λόγω της άμεσης και της έμεσης αλλαγής χρήσης γης. Είναι λοιπόν ευαίσθητο το θέμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζει μερικώς η πρόταση της Κομισιόν, αλλά θα μπορούσε να πάει και πιο μακριά. Το ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι γιατί δεν πρόσθεσε έμεση αλλαγή χρήση γη στα κριτήρια ε, εφορία ω έμεσο τρόπο αντιμετώπιση του προβλήματο. Και δεύτερον, ενώ υποστηρίζω το ανώτατο όριο του 5 ή 10% σε θέματα μεταφορών, μήπω θα έπρεπε να είναι υψηλότερο, ίσως κάποιο απόλυτο ανώτατο όριο όσον αφορά το ποσό χρήση γη για βιοκαύσιμα αλλά και στόχο κίνησης προς το 0% χρήσης βιοκαυσίμων που βασίζονται σε παραγωγή γης ε, και μετά όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων με τα κριτήρια εφορίας που διατυπώνονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε απλά να βασιστείτε ε, στις εκθέσεις των οικονομικών φορέων. Ε, τι ακριβώ προτίθεται να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Μπελαγκλατσέλντερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ε, ότι υπάρχουν διάφοροι στόχοι μέσω της χρήσης βιοκαυσίμων. Ο ένας είναι μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και ο άλλος στόχος όμως είναι η μείωση της ε, ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Προφανώς η παρούσα πρόταση δεν εξυπηρετεί αυτό το δεύτερο στόχο, διότι αν κοιτάξετε την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ευρώπη, τότε δυστυχώς παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο ντίζελ από ό,τι θα έπρεπε. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται να εισάγουμε πετρέλαιο για να έχουμε αρκετό ντίζελ. Ωστόσο, η βενζίνη που αποκτάμε μέσω αυτής της διαδικασίας είναι περιττή, έχουμε περίσσια βενζίνης και χρειάζεται, υποχρεούμαστε να την εξάγουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε χαμηλές τιμές. Αν λοιπόν χαμηλώσουμε, μειώσουμε την παραγωγή βιοκαυσίμου, ε, δίζελ μάλλον όπως λέγεται στην πρόταση, τότε σαφώς θα αυξηθεί η ενεργειακή μας εξάρτηση στην Ευρώπη. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι αυτός ο συντελεστής ε, Άιλακ που αναφέρεται. Δεν υποστηρίζεται με επιστημονικά τεκμήρια. Η νομοθεσία μιλάει για εκτιμήσεις πολύ συχνά στο κείμενό τη, το οποίο σημαίνει ότι εκείνοι που συντάσσουν την νομοθεσία δεν είναι βέβαιοι όσον αφορά αυτή τη μεθοδολογία, κατά πόσο είναι ακριβή ή όχι. Ε, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε περιορισμό του διεθνούς εμπορίου την εισαγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ δεν θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη αυτή η πρόταση. Πολλές ε, ε, συναντήσει οργανώθηκαν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου Βραζιλιάνοι ε, συνεργάτες ανέφεραν ότι μελετούν την πρόταση για να δουν πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό στο επίπεδο ΠΟΕ και πιστεύω ότι φυσικά θα έχουν όλες τις ευκαιρίες για να το επιτύχουν, διότι κοιτάζοντας τους κανόνες του ΠΟΕ δεν υπάρχουν κανόνες που να επιτρέπουν τέτοιους περιορισμούς. Το τρίτο που θα ήθελα να πω αφορά την ερώτηση της πρώτης και των βιοκαυσίμων πρώτης και δεύτερης γενιάς. Είναι σαφές, επαρκώς κατά την απόψή μου, ότι το θέμα εδώ δεν είναι αν τα βιοκαύσιμα είναι πρώτη ή δεύτερη γενιά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτή η περικοπή. Η πρόταση που έχουμε εδώ μπροστά μας δεν μας βοηθάει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πλέουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα και πάμε να δοκιμάσουμε μεθόδους που δεν έχουν δοκιμαστεί. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουμε σε διέξοδο επειδή προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά ως βιοκαύσιμα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει νόημα δηλαδή να κατασκευάζουμε βιοκαύσιμα από ξύλο, διότι το ξύλο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση. Εγώ έχω ε, μια θερμαστραβιομάζας... Ε, ένα τα βιομάζα στο σπίτι και επιτυχάνουν αποτελεσματικότητα 95% με αυτό. Αλλά δεν πρόκειται να επιτυχούμε αποτελεσματικότητα 95% σε περίπτωση που παράγουμε βιοκαύσιμα από ξύλο. Δεν αποτελεί λοιπόν σωστό κίνητρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει και για τα άχυρα και για κοπριά και για τα λοιπά υλικά που αναφέρονται στη λίστα ως βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Περαιτέρω θέτουμε σε κίνδυνο το στόχο μας του 10% όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Και η τέταρτη παρατηρήση που ήθελα να κάνω κύριε Πρόεδρε είναι ότι δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν υπάρχει κίνητρα για ηλεκτρικές μεταφορές παρά ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πραγματικό η πραγματική νέα τεχνολογία που θα μας οδηγήσει κάπου αλλού. Την υποστηρίζει με 2 δισεκατομμύρια δολάρια ε, η τις μεταφορές αυτές τις ηλεκτρικές. Με 2 δισεκατομμύρια ευρώ υποστηρίζονται στη Γερμανία. Εκχωρήθηκε αυτό το ποσό για τον ίδιο στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει. Να, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ε, υποστηρίξουμε τις ηλεκτρικές μεταφορές διότι αυτό θα μας οδηγούσε πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από την Επιτροπή είναι κανείς εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα τα θέματα που τέθηκαν. Δεν μπορούσαν να παρίστανται αυτή τη στιγμή συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Θα τους ε, δώσουμε τις ερωτήσεις που έγιναν και θα πάρετε τις απαντήσεις. Απλώς μια διευκρίνηση να κάνω. Παρά το γεγονό ότι το κριτήριο της αηφορίας εφαρμόζεται στα βιοκαύσιμα, υπάρχουν και κάποια θέματα μη τήρησης αυτών των κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να καθορίσει ποια βιοκαύσιμα θα υπολογιστούν ώστε να μπορέσουν να φτάσουμε στα κατόφλια των ε, ε χρησιμοποίηση στα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστούμε. Χρειαζόμαστε αυτή την διευκρίνηση. Ο Μπερτ Λάγκια, εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σύντομα όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν ξέρω, δεν κολλάνε εδώ πέρα σε αυτή την οδηγία. Έχουμε μία πρόταση για την υποδομή για τα εναλλακτικά οχήματα. Και ε, εδώ πέρα ασχολούμαστε με τα βιοκαύσιμα όπως είπα. Είπατε, μου δώσατε αρκετά ερεθίσματα, πρέπει να τα συζητήσουμε λεπτομερώς όταν θα υποβληθούν οι τροπολογίες, αλλά εμένα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των εισαγόμενων βιοκαυσίμων. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τα εισαγόμενα από τα εγχώρια. Και δεν είναι δυνατόν, όπως είπα, να ισχύσει η κατάσταση η οποία ε, υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά. Ολοκληρώνεται και η συζήτηση αυτού του θέματος. Χρονοδιάγραμμα. 24-25 Απριλίου στην επόμενη συνάντηση συζητηθεί το σχέδιο γνωμοδότησης. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της φορτωμένης ημέρας. Φτάνουμε στο τελευταίο θέμα μας, το 17. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματική διεκτησία και συγγενικών δικαιωμάτων χωρί ιδιαίτερη πολλαπλή ελαφρική ισχύω όσον αφορά τα μουσικά έργα για επιγραμμικέ χρήσει στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για νομοθετικού περιεχομένου φάκελο. Υπεύθυνη τη ουσία είναι η νομική επιτροπή. Η συγητής μας είναι ο Χέλμουτ Σόλτς. Κυρίως για τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε αργήσει λίγο. Ε, το θέμα αυτό δεν το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας. Ε, η Επιτροπή Αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και θα έπρεπε να δούμε το θέμα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια με το σχέδιο έκθεσης. Ας κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Ήρθε και η Κομισιόν, συμμετείχε στη συζήτηση. Είχαμε συζητήσει με του ενδιαφερόμενου. Εμείς είπαμε πως η Επιτροπή μας το έμαθε αργά, τελευταία στιγμή. Ε, το συζητούσα ένα χρόνο ήδη στην ε, ε, Επιτροπή Γιούρη. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα λοιπόν που θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα να πω πως ε, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και καλωσορίζω το ότι ξανασυζητάμε το όλο θέμα από την Επιτροπή διορθώνοντας κατά κάποιο τρόπο τον κανονισμό του 2005. Γιατί θεωρώ πως υπάρχει πραγματικά ανάγκη να διασφαλίσουμε τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων που ε, πρέπει νομίζω να περάσει τώρα από το αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. Έχουμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο ρόλο δεδομένου του ότι το ίντερνετ δεν σέβεται σύνορα. Τα προστατευόμενα έργα πλέον μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου, οπότε η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πρέπει να επανεξεταστεί και οι ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο δημιουργούν και κάποιες πτυχές, δηλαδή δεν μπορούμε μόνο να κοιτάμε τα της εσωτερικής αγοράς και να αποκλείουμε την παγκόσμια πτυχή του θέματος. Αυτό σημαίνει πως αυτό το διαδίκτυο, όπως λέγεται, επηρεάζει την άσκηση ε, και την διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών και Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα μία πτυχή του καταναλωτή. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της εταιρεία που συλλέγει τα δικαιώματα, του κατόχρων εταιρεια που συλλεγει τα δικαιωματα του κατόχων δικαιωματων και του συμφέροντος του καταναλωτή και αυτών που απλά είναι ε, καλλιτέχνες ή πολίτες και θέλουν να συνεισφέρουν μέσω του διαδικτύου και να μοιράσουν ε, την παραγωγή τους αυτή. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θα πρέπει να έχουμε πολυμερή αδειοδότηση και αποτελεσματικές κυρώσεις σε διασυνοριακές συναλλαγές και αυτό αναφέρεται κυρίως στον τελείο 3 και 4 όπου θα πρότεινα ως εισηγητής να επικεντρωθούμε και να εστιαστούμε ως ε, Επιτροπή. Επίσης, να ψήσω την προσοχή σας στο ότι ε, υπάρχει δεν υπάρχει ένα γενικό ε, δικαστήριο για τα πνευματικά δικαιώματα και στις 27 ε, χώρες. Οπότε τα πράγματα αντιμετωπίζονται διαφορετικά και ε, δεν ξέρω αν είναι λογικό το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τη διεθνή σκοπιά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί υπήρχε ήδη μια πρόταση από το Spotify για να συσταθεί ένα δικαστήριο με ε, πολυεδαφική αρμοδιότητα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εταιρείε ε, της συλλογική διαχείρισης των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Διασφαλίζοντας, όπως είπαμε, τα δικαιώματα ε, και τη διάθεση του περιεχομένου στα διαφορετικά και να ε, υπάρξει μια πολυεδαφική αδειοδότηση. Ταυτόχρονα Ταυτόχρονα οι ε, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί βρίσκονται σε διαφορετική θέση π.χ. στην Σκανδιναβία ε, σε σχέση με την ε, Νότια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη. Και για το θέμα αυτό θέλω να τονίσω και τη σημασία του άρθρου 5 παράγραφος 6 που υπάρχουν ρητρες opt opt-in και opt-out. Και αναφερόμαστε σε δικαιώματα και υποχρεώσεις έξω ευρωπαϊκών προμηθευτών. Επίσης να τονίσω πως ε, στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου υπήρχαν ήδη συζητήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι ένας ε, διεθνής οργανισμός που έχει ήδη υπογράψει μία σχετική συνθήκη για την παροχή τεχνικής αρρωγής σε αναψώμενες χώρες για να δημιουργήσουν τέτοιες εταιρείες. και βεβαίω. Επειδή εμεί είμαστε πρωτοπόροι, πρέπει να βοηθήσουμε και άλλε χώρε προ αυτή την κατεύθυνση. Too long. Uh, I want also to stress that strengthening of uh, protection offered to right holders, so that, for example. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η προστασία του κατόχου του δικαιώματος για να έχει δικαίωμα να διακόψει την σύμβασή του με την Εταιρεία Συλλογής Δικαιωμάτων εντός τριών και όχι έξι μηνών. Βεβαίω υπάρχουν και άλλες επιτροπές που επηρεάζονται από την οδηγία αυτή, αλλά δεν μπορούμε να ε, μην την κρίνουμε και από τη σκοπιά του διεθνούς εμπορίου. Και να τονίσω ένα σημαντικό ζήτημα. το οποίο είχα ήδη την ευκαιρία να συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συνθετών και Τραγουδοποιών που λένε πως εάν πάμε στις ΙΠΑ θα δούμε πως έχουμε δύο διαφορετικές πρακτικές. Δεν υπάρχουν εταιρείε συλλογικής διαχείρισης εκεί πέρα και ενώ προσπαθούμε να τις διασφαλίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εμπλεκόμενο διαδικασία θα αντιμετωπίσουμε την αμερικανική πρακτική όπου υπάρχουν άμεσες αδειοδοτήσεις από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει ένα ανάλογο κεφάλαιο στις διεθνείς συνθήκες που να επισημαίνει τις διαφορετικές πρακτικές που επικρατούν στη ΣΥΠΑ. Οπότε Προς αυτή την κατεύθυνση θα πάει η γνωμοδότησή μου. Reflecting of all aspects uh, of this very modern uh, theme uh, and so that our committee is contributing to a approach of the European. Βεβαίως, uh, όπως είπα, πρέπει να έχουμε αυτή τη συλλογική αντιμετώπιση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Helmut Scholl. Πρέπει να πω ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκανα δεν έχουν και μεγάλη σχέση με αυτό τον κανονισμό. Θα μας πούνε πάλι ότι μπαίνουμε στα χωράφια της υπεύθυνσης της ουσίας της Τζούρι. Ο Κρίστοφερ Φιέλνερ, σκιώδης συγγετής για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Διότι πρέπει να εγώ γρήγορα γιατί έχω μια συζήτηση στο νορβηγικό ραδιόφωνο με τον νορβηγικό Υπουργό Γεωργίας ε, για το θέμα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω νορβηγικά, λέει ο πρόεδρο. Μακάρι να μπορούσα και εγώ, λέει ο κύριο Χέλνερ. Αυτό είναι το κύριο μου πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Μου άρεσαν πολλά από αυτά που άκουσα για αυτή τη γνωμοδότηση που όλοι αναμένουμε και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Ε, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα τη μουσική και θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση και πολύ σημαντική. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Spotify και μου φάνηκε τόσο παράξενο που μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στο Χόλμη και μετά ερχόμουν στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω άλλα στη Γαλλία πριν, δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και τώρα μπορώ. Είναι πολύ παράξενο. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει να δημιουργήσουμε κάποιε σωστέ επιλογέ νομικά για το μέλλον και να απλοποιήσουμε τι διαδικασίε. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό, κοιτώντα αυτό εδώ. Και ένα από τα πράγματα που είδα, που έχει διεθνή διάσταση, που είδα στο αυτό το σχέδιο του κ. Σιγητή τη Επιτροπή Γιούρη, είναι ότι μιλάει για την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ανάγκη ρύθμιση αυτή τη ποικιλομορφία. Ε, αυτό θα έχει συνέπειε στο διεθνέ εμπόριο πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί τρόποι αντιμετώπισης της ε, πολιτιστικής πληροφο... Ε, πολυμορφίας, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αδειοδότηση, διότι στο που έχουμε κόκκινες, ε, κίτρινες, λευκές βίβλους, υπάρχουν Μπορούμε να υποστηρίζουμε τον πολιτισμό, αλλά η αδιαδότηση μπορεί να είναι πολύ στο κόκκινο από αψή ΠΟΕ θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη μουσική όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεύτερον, ε, κοιτώντα αυτή την ιδέα του One Stop Shop, του ενίου σημείου εξυπηρέτηση, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο και να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί διεθνώ. Δηλαδή δεν θα είναι μια σημείο εξυπηρετής μόνο για του Ευρωπαίου μόνο από ευρωπαϊκή άποψη. Δυστυχώς πρέπει να φύγω, αλλά θα σας παρακολουθώ και όταν θα λείπω. Και θα αναμένω τις μελλοντικές συζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μα όρια και πρέπει να σας πω ότι οι διερμηνεί θα χρειαστεί να μας εγκαταλείψουν και έχουν και δίκιο. Τους ευχαριστώ λοιπόν που μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω. Από τώρα και στο εξή θα συνεχίσουμε χωρίς δερμηνία στα αγγλικά. Mrs. Martin Abreu, Diabreu. Thank you, Mr. Chair, and thanks for uh, giving the floor to the Commission. And thank you for Mr. Schultz